Πρόκειται για ερώτηση προφορική προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του κεφαλαίου 1 των Βρυξελών 1 σχετικά με τη συμπερίληψη των συμφώνων συμβίωσης. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Γκέπχαρτ. Εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε και κύριοι, στι 18 Ιανουαρίου ενεστώτος έτους πήραμε μια πολύ καλή απόφαση σε μια πολύ καλή βάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ε, πλήρη αναγνώριση και εκτέλεση ε, ζητημάτων σχετικών με ε, το γάμο και την ευθύνη των γονέων. Χάρηκα πάρα πολύ για αυτή την πρόταση γιατί είχαν υιοθετηθεί και δικές μου προτάσεις από παλαιότερη έκθεση. Και είναι καλή νομοθεσία. Έχουμε περισσότερη ασφάλεια δικαίου, ταχύτερες αποφάσεις θα λαμβάνονται και για μας είναι πολύ σημαντικό ιδιαίτερα όταν τίθεται θέμα επιμέλειας τέκνων. Πλην όμως η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει μια πολύ μεγάλη ατέλεια, γιατί ισχύει μόνο για ε, παντρεμένα ζευγάρια. Οι καταχωρισμένες μορφές συμβίωσης εξαιρούνται. Αυτό είναι τελείως αφόρητο, απαράδεκτο, κύριε Επίτροπε, διότι όλο και περισσότερο έχουμε μορφές συμβίωσης καταχωρισμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτός γάμου. Όλο και λιγότεροι άνθρωποι παντρεύονται η κοινωνία αλλάζει, ε, ο τρόπος συμβίωσης και ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εθελοτυφλεί. Για ποιο λόγο, δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Ερμητικά κλειστά τα μάτια σας. Είναι αναδιατύπωση αυτή τη οδηγία και για του πολίτε που μα ακούνε και δεν ξέρουν τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να αλλάξει μόνο εκείνα τα άρθρα τα οποία έχει τροποποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή τροπολογίε απαγορεύεται να καταθέσουμε για το πεδίο εφαρμογή. Δεν είχαμε τη δυνατότητα αυτή ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να φροντίσουμε να επεκταθεί η ισχύ αυτού του νόμου και στι καταχωρισμένε μορφέ συμβίωση. Και για μένα αυτό είναι πάρα πολύ οπισθοδρομικό, πάρα πολύ από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κοιτάξτε λίγο τα ίδια σα τα αριθμητικά στοιχεία και τη Eurostat, που είναι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπηρεσία. Εσεί τα συλλέγετε ο κόσμος παντρεύεται όλο και λιγότερο. Οι άνθρωποι συμβιούν σε μορφές καταχωρισμένης συμβίωσης. Για ποιο λόγο οι άνθρωποι αυτοί που δεν παντρεύονται αλλά επιλέγουν αυτή τη συμβίωση να μην έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους άλλους και τις ίδιες δυνατότητες με τα παντρεμένα ζευγάρια. Για ποιο λόγο οι άνθρωποι σε 19 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορούν ε, να έχουν αυτά ε, τα δικαιώματα και μάλιστα να υιοθετούν πολλές φορές γιατί αποκλείονται από τη συγκεκριμένη νομοθεσία που είναι πολύ καλή. Ερωτώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ποιο λόγο συμβαίνουν όλα αυτά, γιατί έχετε εξαιρέσει τις καταχωρισμένες μορφές συμβίωσης στον κανονισμό Βρυξέλλες 2α. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θεωρεί ότι πρέπει να ρυθμιστεί αυτό για τα συγκεκριμένα ζευγάρια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλείοντας αυτά τα ζευγάρια και αυτές τις μορφές συμβίωσης δεν βλέπει ότι γίνεται διάκριση και βεβαίως γίνεται διάκριση λέω εγώ και εσείς κατά τα άλλα είστε θεματοφύλακα των συνθήκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις συνθήκες η μη διάκριση είναι μία από τις μεγάλες αξίες και αρχές τις οποίες πάντα συζητούμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να διορθώσει αυτή την ε, ε, αμέλεια στο προσεχές διάστημα αν όχι γιατί και αν ναι πότε. Γιατί και αυτό είναι ένα κομβικό ερώτημα. Είναι ε, μεγάλη ευκαιρία που χάθηκε δυστυχώς και περιμένω να ακούσω πολλοί τους συναδέλφους μου από τη δεξιά πτέρυγα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μέχρι τελευταία στιγμή προσπάθησαν να εμποδίσουν να έρθει αυτή η προφορική ερώτηση στην Ολομέλεια προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό το βρίσκω ε, αφόρητο και απαράδεκτο. Γιατί δεν δέχεστε οι άνθρωποι αυτοί που επιλέγουν να ε, καταχωριστούν σε μια μορφή συμβίωση που δεν είναι ε, ε, γάμος να έχουν τα ίδια δικαιώματα. Κύριε Επίτροπε, εσείς στην ψηφιοποίηση θεωρείστε από τους πιο προοδευτικούς και ανοιχτού στο μυαλό που λέει ότι ναι βεβαίως θα πρέπει η κοινωνία μας να αντικατοπτρίζεται στην νομοθεσία μας. Περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω τι θα απαντήσετε σε αυτή την προφορική ερώτηση. Διότι αυτά που ζούμε εμείς εδώ είναι τελείως οπισθοδρομικά και απαράδεκτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο αρμόδιος ε, αντιπρόεδρος, ο κ. Σάντσιπ, θα απαντήσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητά μέλη. Θέλω να σας ευχαριστήσω γενικά που θέσατε το θέμα αυτό των συμφώνων συμβίωσης στα πλαίσια του ΡΙΚΑΣΤ ε, ε, του κανονισμού Βρυξέλλες 2α. Η πρόταση αυτή διευκολύνει την επίλυση νομικών θεμάτων και προβλημάτων σε επίπεδο οικογενειακού δικαίου και σε επίπεδο προστασίας των παιδιών. Η πρότασή μας προσπαθεί να καλύψει τις δυσκολίες που υπάρχουν σε σχέση με θέματα γονικής ευθύνης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ασχοληθεί με τα θέματα αυτά στο παρελθόν και απαιτείται πλέον να αναλάβουμε δράση. Όπως έχει παρατηρήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχουμε προτείνει αλλαγές στις ρυθμίσεις που έχουν σχέση με τον γάμο και δεν έχουμε διευρύνει την δυνατότητα του ζεύγους να επιλέγει την νομική δικαιοδοσία ή ε, δεν έχουμε συμπεριλάβει την προβληματική των ε, ε, συμφώνων συμβίωσης ή των ομόφυλων ζευγαριών. Εμείς δεν είχαμε τις, την απαιτούμενη τεκμηρίωση που να επισημοποιεί, αν θέλετε, το επίγον του θέματος αυτό. Αξιολογήσαμε ότι δεν είναι η σωστή στιγμή αλλαγή των συγκεκριμένων κανόνων βασικός στόχος των Βρυξελών 2α είναι η βελτίωση των τέκνων που αντιμετωπίζουν περίπλοκες και δύσκολες καταστάσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί επιγόντως. Εδώ εκφράζω την ικανοποίησή μου διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή ε, θέλουν να αποτρέψουν τα παιδιά να παραμείνουν ως όμοιροι μακροπρόθεσμων κατά τα άλλα δικαστικών διαδικασιών. Θέλουμε να απλουστεύσουμε τις δικαστικές διαδικασίες μειώνοντας και το κόστος αλλά και τον χρόνο, το μήκος τους. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπίπτουν στην δυνατότητα παροχής ε, του ιδίου επίπεδου προστασίας σε όλα τα παιδιά. Να υπογραμμίσω ότι στην δική μας πρόταση διευκρινίσαμε ότι η σωστή προστασία των παιδιών καλύπτει το σύνολο των παιδιών ανεξαρτήτως ε, του καθεστώτος ε, των γονέων τους ανεξαρτήτως του εάν είναι νηφευμένοι ή αν είναι στο εσωτερικό είναι νυφευμένοι ή αν είναι σε, ε, στο εσωτερικό ενός συμφώνου συμβίωσης. Και θυμίζω επίσης ότι στο Συμβούλιο απαιτείται ομοφωνία για όλα τα θέματα αυτά. Συνεπώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις έτσι ώστε να υπάρξει μια σωστή ε, κατάληξη στη διαδικασία αυτή προς όφελος των νέων παιδιών. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Να δώσω το λόγο στην κυρία Σταράς Φερακούτ για δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, ο βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να διατηρήσει το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό να μπορεί να υπάρχει συνεργασία σε δικαστικό επίπεδο, κυρίως όσον αφορά τα οικογενειακά θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό ακριβώς και μαζί με τον εισηγητή παρουσιάσαμε ε, μία αναδιαμόρφωση όλου αυτού του οικογενειακού δικαίου που θα αποτελούσε και ένα βήμα ε, προς το μέλλον για να υπάρχει ασφάλεια δικαίου, για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις, σύγχυση και να αποτελέσει και τον ακρογωνίο λίθο αυτής της δικαστικής συνεργασία. Υπήρχαν ομοιόμορφες διαδικασίες όσον αφορά το χωρισμό, το διαζύγιο, ε, τα αγωνικά θέματα ε, και την αντιμετώπιση διασυνοριακών περιπτώσεων, οι οποίες όπως γνωρίζετε αυξάνονται συνεχώς. Θα υπήρχε έτσι ελεύθερη κυκλοφορία αποφάσεων, δικαστικών αποφάσεων, εγγράφων και φυσικά υπάρχουν και ε, θέματα τα οποία πάντα είναι εις βάρος των ανηλίκων που ήταν και το βασικό αντικείμενο αυτής της πρότασης. Το είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που έχουν ρυθμίσει τα σχετικά θέματα, αλλά υπάρχουν και άλλε χώρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχουν ρυθμίσει και είναι μια πραγματικότητα και πιο σημαντική. Υπάρχουν παιδιά τα οποία γεννιούνται από ζεύγη, τα οποία δεν είναι παντρεμένα και υπάρχουν και πολλά ε, ζευγάρια τα οποία έχουν σύμφωνο συμβίωση. Γι' αυτό ακριβώ ε, και θεωρούμε ότι θα πρέπει ε, να λάβουμε υπόψη αυτή την πραγματικότητα. η Επιτροπή θεωρεί ότι θα θέσει σε κίνδυνο τη συμφωνία, ενώ στην πραγματικότητα ο στόχο πάντα είναι να προστατεύσουμε του ανηλίκου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βιώτη για 1,5 λεπτό. Να σας ευχαριστήσω Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο. Η ερώτηση αυτή έχει ειδικό βάρος θα έλεγα για πολλούς Ευρωπαίους πολίτες. Οι δυνατότητες τις οποίες έχει βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση στο να παρεμβαίνει σε θέματα αστικού δικαίου είναι λίγες. Ε, οι Βρυξέλλες 2α επιτρέπουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις στον τομέα των, της γονικής ευθύνης κτλ. Στο εσωτερικό του κανονισμού αυτού λοιπόν, Βρυξέλλες 2, οι μη νυφευμένοι αυτοί οι οποίοι ζουν σε σύμφωνο συμβίωσης, όπως επίσης και τα ζεύγη τα ομόφυλα, ε, νομίζω θέτουν οι κατηγορίες αυτές ένα δεοντολογικό πρόβλημα. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε και τους πολίτες αυτούς και κυρίως να προστατεύσουμε τα παιδιά τα οποία είναι στο εσωτερικό αυτών των, ε, των, των ε, ζευγών. Συνεπώς λοιπόν είναι πλέον, έχει φτάσει η ώρα για να καταπολεμήσουμε αυτές τις διακρίσεις. Μιλάμε για κράτος δικαίου πολύ συχνά, επανειλημμένα. Είναι λοιπόν μια περίπτωση εδώ που η Ευρώπη μπορεί να κάνει κάτι. Είπατε Επίτροπε ότι δεν έχει φτάσει η στιγμή για να συζητήσουμε αυτήν την αναγνώριση. Κοιτάξτε, ε, η σωστή στιγμή για την αναγνώριση ενός δικαιώματος είναι πάντα το χθες. Γιούρεκ. Ευχαριστώ. Η οικογένεια η οποία μπορεί μερικές φορές να βασίζεται σε ένα νομικό πλαίσιο συμβίωσης, σε σύμφωνο συμβίωσης, είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει και την κοινωνία μας σήμερα. Πάντως δεν θα πρέπει την παραδοσιακή μορφή της οικογένειας να την θέσουμε στο ίδιο επίπεδο με άλλου είδους σχέσεις οι οποίες είναι αυστηρά θα έλεγα όχι κοινωνικού αλλά ιδιωτικού χαρακτήρα. Έτσι θα διασφαλίσουμε το μέλλον για τις κοινωνίες μας. Και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην ξεκινήσει ε, να λαμβάνει μέτρα πολιτικά εις βάρος των χωρών οι οποίες είναι πιστές στις βασικές αλήθειες της κοινωνίας μας. Οι αποφάσεις οι οποίες ε, λαμβάνονται μερικές φορές ε, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι συμβατές ε, με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την υποχρέωση να μην παρεμβαίνει σε οικογενειακά θέματα και πρέπει να τηρήσει το λόγο της. Η κυρία Χάουταλα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Αντιπρόεδρε, θα συμφωνήσω με αυτά τα οποία είπε ο συνάδελφος Βιώτη ότι έχει φτάσει η στιγμή να κάνουμε πραγματικότητα αυτά τα οποία πρεσβεύουμε. Ανησυχούμε για το κράτος δικαίου, ανησυχούμε για τα δικαιώματα των πολιτών και δεν πρέπει να χάνουμε πλέον χρόνο. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, χρησιμοποιώντας την τεχνική του recast της αναδιατύπωσης έχει δέσει τα χέρια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το κείμενο λοιπόν το ανανεωμένο υποτίθεται ότι πρέπει να βοηθήσει την ταχεία λήψης αποφάσεων η οποία είναι ίδια εδώ και 15 χρόνια. Καιρός είναι να εξυγχρονιστεί και στις νέες μορφές οικογενειακής συμβίωσης. Πριν 15 χρόνια δεν ήταν αναγνωρισμένες οι μορφές αυτές, τώρα εν πολλής είναι, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη λοιπόν και τα συμφέροντα αυτών που βρίσκονται σε σύμφωνα συμβίωσης. Ευχαριστώ. Γκούτελαντ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αν είναι φιλική προς τα παιδιά, αυτό είναι κάτι καλό για όλους εμάς. Η οικογένεια στην Ευρώπη είναι πολύ σημαντική. Θα πρέπει τα παιδιά να μεγαλώνουν με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος που συνδέει τους γονείς τους. Όλο και περισσότερα παιδιά γεννιούνται εκτός γάμου. Και μάλιστα οι γονείς τους ζουν σε διαφορετικές χώρες. Όλο και περισσότερα παιδιά γεννιούνται από, παιδιά, από ε, γονείς με σύμφωνο συμβίωσης που δεν είναι παντρεμένοι. Είναι πραγματικά κρίμα να βλέπουμε με ποιο τρόπο ε, κάποια πτέρυγες εδώ του Κοινοβουλίου αντιτίθενται ε, σε κάποια προοδευτικά μέτρα. Ενώ 19 κράτη-μέλη, μεταξύ αυτών και η Σουηδία, προβλέπουν αυτά τα σύμφωνα συμβίωσης. Ο γάμος πολλές φορές και σε πολλές ε, χώρες αφορά ε, ζευγάρια του αντίθετου φύλου. Ε, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά στην Ευρώπη, των οποίων το νομικό καθεστώς είναι μετέωρο. Τι θα κάνουμε με τα σύμφωνα συμβίωσης, πώς θα προστατεύουμε τα παιδιά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι πιστεύει και τι προθέσεις έχει. Θα επεκτείνει το πεδίο εφαρμογή. κυρία Ράιντκε, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητέ Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρέπει να πω ότι δυστυχώς, δυστυχώς και το τονίζω ακόμα σήμερα, δεν έχουν αναγνωρίσει ε, ε, τα, ε, το γάμο στα μόφυλα ζευγάρια όλες οι χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα πλήρη ισότητα και έτσι τα σύμφωνα συμβίωσης και οι καταχωρισμένε μορφές συμβίωσης θα πρέπει να εξισώνονται με το γάμο όσο δεν αναγνωρίζεται παντού ο γάμο. Κύριε Επίτροπε, μα φέρατε διάφορα επιχειρήματα. Όλα αυτά δεν είναι αντίθετα με τη συμπερίληψη των συμφώνων συμβίωσης στην νομοθεσία αυτή. Το μοναδικό επιχείρημα που βλέπω αυτή τη στιγμή να είναι επιτάπητο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει πλάτε σε δεξιέ κυβερνήσει που δεν θέλουν αυτά τα σύμφωνα συμβίωση και τα ομόφυλα ζευγάρια. Εμεί είμαστε υπέρ του κράτου δικαίου, ε, τη ισότητα και τη ελευθερία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα υπερασπιζόμαστε. Ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να το κάνει αυτό. Διότι όλοι οι πολίτες αξίζουν να έχουν τα ίδια δικαιώματα. Ευχαριστούμε. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Και τώρα ξεκινάμε τη διαδικασία Catch the Eye. Έχουμε τέσσερις συναδέλφους. Η κυρία Μαριάννα Πετήρ έχει πρώτο λόγο. Μικρόφωνο παρακαλώ. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να τροποποιήσει εν μέρη τον κανονισμό ε, είναι ευπρόσδεκτη από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι είναι προφανές ότι το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για το οικογενειακό δίκαιο δεν ρυθμίζει τα ευαίσθητα ζητήματα με ικανοποιητικό τρόπο. Επειδή ο κανονισμός Βρυξέλλες 2 καθορίζει την αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων, το Συμβούλιο δεν θα μπορεί ε, να εκρίνει την παράταση του πεδίου εφαρμογής ε, και για τις καταχωρημένες ε, και για την καταχωρημένη συμβίωση, διότι δεν υπάρχει στο νομικό σύστημα κάποιων κρατών μελών. Θα έχει άμεση συνέπειες για την εθνική νομοθεσία και τις αρχές του γάμου και της οικογένειας και παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας. Ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην επεκτείνει το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού γιατί θα δημιουργήσει διτές καταστάσεις και θα διευρύνει το χάσμα μεταξύ των κρατών που έχουν καταχωρισμένη συμβίωση και αυτών που δεν διαθέτουν. Ε, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα θέματα της τεκνοθεσίας. Θα πρέπει λοιπόν να εναρμονίσουμε τα νομικά μας συστήματα. Δεν χρειάζεται διαιρέσεις και πολιτικές πιέσεις προς τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ η κυρία Γκραπίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Γκέπχαρτ, η οποία παρουσίασε πολύ ισχυρά επιχειρήματα για τη λύση αυτού του προβλήματος, ε, για το οποίο περιμένουμε απάντηση. Τα πράγματα ε, εξελίσσονται. Εμεί Εμείς γνωρίζουμε και στη χώρα μου πολλές ε, περιπτώσεις σχέσεων και οικογενειών που έχουν δημιουργήσει νέοι άνθρωποι οι οποίοι δεν παντρεύονται αλλά κάνουν παιδιά. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν δικαιώματα για αυτά τα παιδιά γιατί μετά από 5-10 ε, χρόνια ε, χωρίζουν αυτά τα ζευγάρια και τα παιδιά βρίσκονται σε μια επισφαλή κατάσταση. Κύριε Επίτροπε, επιτρέψτε μου να σας κάνω μια ερώτηση. Είπατε ότι δεν σκεφτήκατε την τροποποίηση του κανονισμού διότι μετά από τη δημόσια διαβούλευση δεν θεωρήθηκε απαραίτητο. Μήπω θα μπορούσατε να διαβιβάσετε στο Κοινοβούλιο αυτή τη μελέτη πόσε δυνατότητε συμφώνου συμβίωση υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσα σύμφωνα έχουμε, πόσα παιδιά γεννιούνται σε αυτά τα σύμφωνα, ε, πώς δικαιολογείται ότι δεν χρειαζόμαστε αλλαγέ. Ο κύριος Χατζηγεωργίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Κέπχαρτ, διότι έφερε στο Κοινοβούλιο ένα πάρα πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Και είναι πραγματικά, θα το πω με έκπληξη, που άκουσα ότι δεν ρυθμίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση το, νομικό στάτους των παιδιών ε, που βρίσκονται ε, μέσα σε ένα σύμφωνο συμβίωσης των γονιών τους. Αλλά μου προκάλεσε πολύ μεγαλύτερη έκπληξη η απάντηση της Επιτροπής που οφείλω να πω δεν την κατανόησα πλήρως. Ως να έλεγε ο Επίτροπος ότι δεν ισχύει αυτό διότι συμπεριλαμβάνονται και τα παιδιά από σύμφωνο συμβίωση αλλά στη συνέχεια σαν να κάτι άκουσα περί συμφωνίας όλων των κρατών μελών νομίζω ότι αυτό χρειάζεται μια καθαρή διευκρίνηση και δεν χρειάζεται τέλος να επαναλάβω και εγώ ότι χιλιάδες πλέον παιδιά γεννιούνται ε, χωρίς οι γονείς τους να είναι παντρεμένοι με τον καθιερωμένο τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Sorry. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη κύριε Επίτροπε, γνωρίζουμε ότι ούτε σήμερα ούτε το 2015 υπήρχε ομοφωνία στο Συμβούλιο για τον κανονισμό αυτό, για το οικογενειακό δίκαιο και την ε, υποστήριξη των συμφώνων συμβίωσης. Υπάρχουν χώρες αντίθετες προς τις ρυθμίσεις αυτές. Αυτό δεν θα πρέπει να έρχεται σε σύγκρουση ούτε κατά διάνοια με το οικογενειακό δίκαιο της κάθε χώρας. Για ποιο λόγο μας απασχολεί σήμερα αυτό το θέμα και το συζητούμε. Είναι σαφέστατο για να δημιουργηθεί ε, πολιτική πίεση ε, απέναντι στις χώρες αυτές που έχουν κάποια συγκεκριμένη εικόνα για την οικογένεια και δεν υποστηρίζουν τις σύγχρονες τάσεις. Εκπλήσωμαι που βρίσκουν χώρο εδώ τέτοιες συζητήσεις και τέτοια επιχειρήματα. Ο κύριος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει το λόγο παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, χωρίς μικρόφωνο συνεχίζει ο Επίτροπος. Το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και πάλι για τη συνεχή στήριξη στις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και γιατί θέτετε πολύ σημαντικά θέματα για το περιεχόμενο των προτάσεων. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει επαρκές ενδείξεις οι οποίες να δικαιολογούν ε, πρόταση για τροποποίηση των διατάξεων του κανονισμού Βρυξέλλες 2α για τα οικογενειακά θέματα. Ωστόσο, έχουμε εξασφαλίσει ότι όλες οι διατάξεις ε, που στόχο έχουν να βελτιώσουν την προστασία των παιδιών θα εφαρμόζονται ισότιμα για όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από την ε, οικογενειακή κατάσταση ε, της οικογένειας την οποία ζουν. Τα παιδιά βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της μεταρρύθμισης. Ο χωρισμός των γονιών τους είναι αρκετά δύσκολος από μόνος του χρειάζονται διαδικασίες οι οποίες διευκρινίζουν την κατάστασή τους το συντομότερο δυνατόν και λαμβάνουν υπόψη το συμφέρον του παιδιού. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να επιταχύνουμε ε, ιδίω όσον αφορά τις διασυνοριακές υποθέσεις και πρέπει να εφαρμοστούν αυτοί οι νέοι κανόνες πολύ γρήγορα για το καλό των παιδιών. Για να είμαι απόλυτα σαφής, εγώ ήμουνα μεταξύ αυτών που προώθησαν ε, τον πολιτικό γάμο στην Εστονία. Και φυσικά υπερψήφισα το σχετικό νόμο στην Εστονία. Αλλά τώρα ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά μα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, διότι πραγματικά υπάρχουν παιδιά που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση. Και όπω ε, πολύ σωστά ακούσαμε και από μέλη του Κοινοβουλίου ε, και όπω είπα και εγώ στην αρχή, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά χρειάζεται ομοφωνία στο Συμβούλιο. Και ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί αυτή η ομοφωνία εάν επεκτείνουμε την πρόταση και στο Σύμφωνο Συμβίωσης. Γιατί λοιπόν να υποβάλουμε τα παιδιά μας σε μια τόσο δύσκολη δοκιμασία. Αυτό είναι το ερώτημα. Πρέπει βέβαια σίγουρα να ασχοληθούμε με τα θέματα αυτά. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Πρέπει να σεβαστούμε και ε, τους γάμους ομοφιλοφίλων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς κύριε Αντιπρόεδρη. Με αυτό ολοκληρώνεται η συζήτηση και περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο.